Przewodniczący! Good morning, please, colleagues. Take Σας καλημέρα, σας καθίστε συνάδελφοι παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα να πω ότι άρχεται η συνεδρίασή μας και θα περάσουμε στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόσθετο σημείο όσον αφορά την κρίση στην Ευρώπη που οφείλεται στις διαταραχές των, ε, της εναέριας κυκλοφορίας. Πρωτού ξεκινήσουμε θα ήθελα κάποιες πληροφορίες να σας δώσω. Στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων σε σχέση με την κατάσταση αυτή και σε επαφή με τις κοινοβουλευτικές ομάδες θα ήθελα να προτείνω τις εξής αλλαγές όσον αφορά την ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Είναι νέες αλλαγές, νέες τροποποίησεις αυτές. Πρόκειται για τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν, εγκρίθηκαν εχθές Κάνω λόγο για πρόσθετες τροποποίησεις, πρόσθετες αλλαγές λοιπόν. Πρώτα απ' όλα διαγράφουμε τον γύρο ερωτήσεων προς το Συμβούλιο από την ημερησία διάταξη. Το είπε το Συμβούλιο αυτό, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Λόπεθ Γαρδίδο θα πρέπει να φύγει από το Στρασβούργο στη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε την απογευματινή, τον απογευματινό χρόνο ερωτήσεων. Δεύτερον, στην έκθεση Σίλβια Τίτσαου θα αφαιρεθεί από την ημερησία διάταξη όσον αφορά τα κτίρια και καθώς η έκθεση δεν είχε εγκριθεί στην ε, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με τη Δευτέρα. Τρίτον, μια προφορική ερώτηση θα συμπεριληφθεί όσον αφορά την ε, απαγόρευση χρήσεως κάποιων τεχνολογιών στα ορυχεία με την χρήση κιανίου και αυτό μετά τη συζήτηση για τα στοιχεία SWIFT και Passenger Name Records, PNR, στοιχεία ταξιδιωτών σε αέριες μεταφορές. Έτσι λοιπόν θα κλείσει η συνεδρίαση της Τετάρτης ε, στις 7 το βράδυ. Έτσι λοιπόν και πάλι εν συντομία διαγράψαμε εκείνα τα σημεία από την ημερήσια διάταξη της Τετάρτης τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν στην Ολομέλεια. Και σαν αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών η Ολομέλεια της Τετάτης θα σταματήσει, θα τερματιστεί όχι τα μεσάνυχτα, τα αλλά θα τερματιστεί στις 19.00 στις 7 το βράδυ. Αυτά σε σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των ομάδων. Ο κύριος Κρέμερ παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Monsieur Kramer. Ο κύριος Κράμερ, παρακαλώ. No, 396. 396. Εσείς παρακαλώ. Δεν παρίσταστε. Εντάξει, δεν παρίστατε. Ευχαριστούμε. Επιλύθηκε το πρόβλημα. Εξαιρετικά. Ο κύριος Ρούμπιχ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα εγώ να ρωτήσω αν την Πέμπτη θα γίνουν κάποιες συνεδριάσεις ε, στο σώμα κοινοβουλευτικών επιτροπών ή ΣΤΟΑ και άλλων, αν μπορούν να συναντηθούν με διερμηνεί προβλέπονται συνεδριάσει και ομάδε επισκεπτών την Πέμπτη θα, μπορούν, να, μπορούμε να τι υποδεχθούμε την Πέμπτη εδώ. πρόεδρο. ακούστε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα τη ερώτησή σα. Ενημερωτικά λοιπόν προετοιμάζω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα υπογράψω εγώ ίδιος ως πρόεδρος και θα απευθύνεται σε όλα